presidente Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Ανακοινώνω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 733 ψηφίσαντες. Απαιτούμενη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου 374. Ψήφι υπέρ 383. Ψήφι κατά 327. Αποχές 22, άκυρα 1. Με βάση τα αποτελέσματα, η υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια στην κυρία Ούρσλα Φόντε Λάιεν για την εκλογή της να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την άσκηση των καθηκόντων της. Βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 3 του κανονισμού θα ενημερώσω το Συμβούλιο και θα καλέσω το Συμβούλιο και την εκλογήσα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνουν μετά από κοινή συμφωνία τους υποψηφίους ε, επιτρόπους. Θα υπογράψω τώρα την επιστολή κοινοποίησης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. E la consegno, visto che è Και επειδή είναι παρούσα, την ε, παραδίδω στην ε, Πρόεδρο. Κυρία Βοντελάιεν, σας συγχαίρω εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκλογή σας στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξ ονόματος των συναδέλφων, ε, βεβαίως και συγχαρητήρια από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Τώρα ξεκινά ένα πολύ σημαντικό στάδιο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επιλογή των επιτρόπων ε, που όπως γνωρίζετε θα ε, συμμετέχουν σε πολύ ε, διεξοδικές ακροάσεις ε, Ελπίζουμε ότι τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε σήμερα στο ημικύκλιο θα ε, τα συνεχίσουν και οι Επίτροποι ε, στη διάρκεια των ακροάσεων στις αρμόδιες επιτροπές. Ε, τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία μόνο εάν υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Σας δίνω το λόγο για να δώσετε κι εσείς ένα μήνυμα ημικύκλιο. Παρακαλώ. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νιώθω τεράστια τιμή. Ε, είμαι καταθουσιασμένη και σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Η εμπιστοσύνη που μου δείξατε είναι η εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη σε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη, από Ανατολάς προς Δυσμά, από Βορρά προς Νότο. Η εμπιστοσύνη σε μια Ευρώπη που είναι έτοιμη να δώσει τη μάχη της για το μέλλον και όχι να ε, σπαράζεται από ε, αλληλοσκοτομούς. Και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις των καιρών μας. Το Έχω ε, συνέστηση της τεράστιας ευθύρης που βρίσκεται μπροστά μου και των τεράστιων προκλήσεων και το έργο μου ξεκινά τώρα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο σας όλοι, όλους τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποφάσισαν ε, να μου δώσουν την ψήφο τους. Πάντως το μήνυμά μου προς όλους σας είναι ας συνεργαστούμε, ας εργαστούμε όλοι μαζί επικοδομητικά. Γιατί ε, κοινός μας στόχος είναι μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φοντελάιεν. Θα διαβιβάσω τώρα τις επιστολές στο Συμβούλιο και βεβαίως και στον πρόεδρο Ντόναλτ Τούσκ για την απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια. Διακόπτεται η συνεδρίαση για μερικά λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται τη συνεδρίαση. Παρακαλώ καθίστε και αν δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε τι εργασίε, παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε την καλοσύνη, όσοι δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε τις ε, εργασίες, ε, να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τη δήλωση τη Αντιπροέδρου Υπάτης Εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για εξωτερικέ υποθέσει και Πολιτική ασφαλεία για την εφαρμογή της ε, Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Να δώσω αμέσως λοιπόν το λόγο στην ε, Υπάτη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο, την κυρία Μογκερίνη, και επειδή είναι η πρώτη φορά που έχω τη χαρά να ε, προεδρεύω στη διάρκεια τη παρέμβασή σα, να σα συγχαρώ και να σα ευχαριστήσω για τα όσα κάνετε στη διάρκεια τη θητεία αυτή και να σα ευχηθώ ό,τι καλύτερο για του τελευταίου μήνε ε, τη θητεία σα και ό,τι καλύτερο και για το μέλλον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά για μένα και τιμή να ε, είμαι αυτή η οποία ξεκινάει την πρώτη συζήτηση, αν κατάλαβα καλά, της ε, ε νέας ε, Ολομέλειας ε, και είχα και την τιμή να είμαι εδώ στην τελευταία συζήτηση. Θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους για την εκλογή, την επανεκλογή σας και να συγχαρώ φυσικά πρώτα απ' όλα τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την Ούρσουλα έχουμε συνεργαστεί πολύ θετικά τα τελευταία χρόνια και Έχουμε συνεργαστεί κυρίως ε, για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Και είμαι βεβαία ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρεθεί σε καλά χέρια. Ε, από τους τομείς συνεργασίας μας ε, με την Ούρσουλα και άλλους υπουργούς εξωτερικών και υπουργούς άμυνας ε, των κρατών μελών, μερικούς μάλιστα τους βλέπω και τώρα στο ημικύκλιο έχουν γίνει ευρωβουλευτές. Ε, κοινό μα στόχο, ε, μεταξύ άλλων, είναι και αυτή η παγκόσμια στρατηγική που αρχικά σχεδιάσαμε, χαράξαμε και εφαρμόσαμε πριν από τρία χρόνια. Η παγκόσμια στρατηγική ήταν η πηξίδα του έργου μα τα τελευταία ε, τρία χρόνια και μάλιστα την προετοιμάσαμε στο παρελθόν και θα ήθελα να, να ευχαριστήσω και το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη κατά τη χάραξη της στρατηγικής αλλά κυρίως για την εφαρμογή της στην πράξη και μάλιστα η παγκόσμια στρατηγική είναι ε, ο καρπό μια κοινή προσπάθεια, συλλογική προσπάθεια και με τα 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κέριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά και με τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, ε, τα think tanks, την κοινωνία των πολιτών. Ήταν πραγματικά ένα συλλογικό έργο. Και η ευκαιρία επίση να επικεντρωθούμε σε αξίε ε, και κοινά μα ενδιαφέροντα έχουμε κάποιε κοινέ αξίε και ενδιαφέροντα, άσχετα από την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκουμε και άσχετα με την ιδεολογική συζήτηση. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και να εδραιώσουμε το παγκόσμιο μα ρόλο ω παρόχου ασφάλεια στο διεθνέ προσκήνιο και οι μείζονε προκλήσει του καιρού απαιτούν πολυμερεί λύσει. Και συμφωνούμε ότι η Ευρώπη θα έχει βαρύτητα και έχει βαρύτητα και κάνει τη διαφορά στον κόσμο μόνο εφόσον αποφαίνεται ε, και δρά ενιαία, ως ενιαία Ευρώπη και ε, ελπίζω να έχετε δει και την παγκόσμια στρατηγική αλλά και την έκθεση που υπέβαλα το προηγούμενο μήνα στο Συμβουλίο Εξωτερικών Γενικών Υποθέσεων μετά τη συζήτηση του περιεχομένου της έκθεσης ε, στις επιτροπές ΔΕΒΕ και ΑΦΕΤ στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Είχαμε 50 πολύ πυκνές σελίδες επιτευμάτων και πιθανών ε, πρωτοβουλειών για το μέλλον. Και αυτή είναι η παρακαταθήκη που σας αφήνω για τις μελλοντικές σας συζητήσεις για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους μηχανισμούς που ήδη προτείναμε και να διαμορφώσετε τη μελλοντική εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε μόνο όμως τρεις άξονες στην παγκόσμια στρατηγική. Θα ήθελα όμως προς το παρόν να επικεντρωθώ σε αυτά τα τρία σημεία. Ασφάλεια και άμυνα, πολυμέρεια και ιδέα μια πιο κοινή ε, προσπάθεια και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν για την ε, άμυνα και την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον έχει πολιτική βούληση, μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα και καρπού. Μερικέ φορέ, μάλιστα, καταφέραμε πολύ περισσότερα από όσα ελπίζαμε και προσδοκούσαμε. Καταφέραμε να θεσπίσουμε τον μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας, τη μόνιμη διαθρωμένη συνεργασία, το ΠΕΣΚΟ. Μερικοί ήταν πολύ δύσπιστη και καχύποπτη στην αρχή και το συζήτησα και πρώτη φορά στην κοινή ακρόση που είχαμε στις Επιτροπές ΔΕΒΕ και ΑΦΕΤ. Και παρά το σκεπτικισμό, παρά τις αντιστάσεις που υπήρχαν, τα καταφέραμε. Και μάλιστα ήμασταν ακόμη πιο φιλόδοξοι με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και την ε, ετήσια συντονισμένη αξιολόγηση για την άμυνα. Και αυτά δεν είναι μόνο αρχικά και ακρονίμια, είναι πραγματικές αλλαγές στην κοινή πολιτική μας για την ασφάλεια. Και θέλουμε οι άμυνες για την, τα κονδύλια για την άμυνα και οι δαπάνε είναι πιο αποτελεσματικέ και να αναπτύξουμε τι στρατιωτικέ ικανότητε που χρειαζόμαστε στου εθέρε, στη θάλασσα, στον κυβερνοχώρο. Οι διεθνεί μα αποστολέ έχουν καλύτερε ε, δομέ διοίκηση και έχουμε δεσμευθεί να επικεντρωθούμε και στι μη στρατιωτικέ δράσει, τι πολιτικέ δράσει, πολιτική προστασία, που είναι το καμάρι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας και άμυνας είχε κάνει τα πρώτα έμπρακτα βήματα και συγκεκριμένα μετά από πολλές δεκαετίες που ήταν μόνο στα χαρτιά ή ούτε καν στα χαρτιά. Και ταυτόχρονα ενώ ε, ενδυναμώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδυναμώνουμε και την ε, στρατηγική μας και τη συνεργασία μας με, στην ασφάλεια και την άμυνα με τους εταίρους μας όλο τον κόσμο, στο ΝΑΤΟ αλλά και πέραν αυτού. Μάλιστα μόλις επέστρεψα από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Εκεί συνεργαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεργαζόμαστε με τις ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες ήμουν στο Σαχέλ. Εκεί βοηθήσαμε τις ε, πέντε χώρες του Σαχέλ να ιδρύσουν μία ε, πολυεθνική στρατιωτική δύναμη. Θέλουμε να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα την πολυμέρεια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεργάσιμη και πολυμερής ίσχυ εξορισμού. Και αυτό είναι το DNA και το ευρωπαϊκού μα σχεδίου. Είμαστε λοιπόν υπέρ του, της πολυμέρειας και παρά της κρίσης που αντιμετωπίζει και το σύστημα του ΟΗΕ θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο από ποτέ στην πολυμέρεια και μάλιστα αναβαθμίσαμε την ε, οικονομική ε, στήριξη στα Ηνωμένα Έθνη για παράδειγμα ε, σώσαμε από την ε, οικονομική κρίση την ε, Ειδική Υπηρεσία για, το, για την Παλαιστίνη των Ηνωμένων Εθνών. Στηρίζουμε την, το ανθρωπιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και θέλουμε πολυμερείς λύσεις στα πολυάριθμα και δύσκολα προβλήματα των καιρών μας. Οπότε όχι μόνο είμαστε υπέρ τη ε, πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, είμαστε υπέρ τη συμφωνία των Παρισιών για τις κλιματικές αλλαγές, υπέρ των βιώσιμων στόχων ανάπτυξη. θέλουμε μια νέα γενιά δίκαιων ε, εμπορικών συμφωνιών. Και ανέκαθεν προσπαθούσαμε να ενισχύσουμε, να δημιουργήσουμε ένα πολυμερές σύστημα, ακόμη και όταν δεν υπήρχε και μετά τη συζήτηση αυτή θα μιλήσουμε για τη Βενεζουέλα και έχουμε την διεθνή ομάδα επαφής που προωθήσαμε και προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Βενεζουέλα. Επίσης, έχουμε πολυμερή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Αφρικανική Ένωση, ε, τη διάσκεψη των Βρυξελών για την Συρία και επίσης τις συναντήσεις για να τη στηρίξουμε την ειρήνη στο Αφγανιστάν. Έχουμε πολύ άριθμα παραδείγματα της πολυμερούς μας προσέγγισης, πολύ απτά μάλιστα παραδείγματα. Όχι μόνο ήμασταν ανέκαθεν υπέρμαχοι της πολυμέρειας, αλλά προτείναμε και καινοτόμες νεοτεριστικές λύσεις για να την ενισχύσουμε. Και σίγουρα πριν από τρία χρόνια, ε, όταν προτείναμε την παγκόσμια στρατηγική, είχαμε μια ιδέα και νομίζω ότι την έχουμε βελτιώσει κατά πολύ. Και θα ήθελα να, βελτίσω, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί η υποστήριξη και από την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία προκειμένου να βελτιώσουμε την συνοχή και την ε, ε, και το συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μέχρι στιγμής ε, ήμασταν επιτυχημένοι όσο ήμασταν ενωμένοι. Και μια πιο ενωμένη Ευρώπη και συσπηρωμένη δεν είναι μόνο μια επιλογή αρχής ε, όταν ακολουθούμε τα βήματα των ιδρυτών πατέρων και μητέρων. Μια ε, ενωμένη Ευρώπη είναι εγγύηση επιτυχίας. Μόνο μια ενωμένη Ευρώπη θα έχει βαρύτητα σήμερα. γιατί δεν έχουμε μόνο μεγάλες και μικρές χώρες μέλη. Έχουμε ε, κάποιες χώρες που δεν έχουν αντιληφθεί, ακόμη και όταν είναι μεγάλες ε, στις διαστάσεις, ότι είναι μικρές παγκοσμίω. Μόνο ενωμένοι λοιπόν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα ε, συμφέροντα και τι αξίε μα. Και όταν μείνουμε ενωμένοι, θα κάνουμε τη διαφορά. Και μερικέ φορέ η διαφορά είναι ζωτική σημασία, όχι μόνο για μα, αλλά και για του εταίρου μα παγκοσμίω. Αυτά λοιπόν τα χρόνια σημειώσαμε, κατά τη γνώμη μου, θεαματική πρόοδο. Για παράδειγμα, συνδέσαμε τις πολιτικές μας της ασφάλειας και της ανάπτυξης την εσωτερική και εξωτερική πλευρά των δράσεών μας με ένα πιο συντονισμένο έργο εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χάρη στην ομάδα που ιδρύσαμε με τους Ευρωπαίους, την ομάδα για την εξωτερική δράση και μάλιστα ε, κάθε μήνα συνεδριά, συνεδριάζει αυτή την πενταετία και με τα κράτη-μέλη. Έχουμε καλύτερο συντονισμό από ποτέ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κάτι που στο παρελθόν φαινόταν ε, αδύνατο μέχρι πριν από μια τριετία. Ε, πάντως, ε, αυτή η επιτυχία κατέστη δυνατή χάρη στην συλλογική πολιτική βούληση για πρόοδο. Και θα ήθελα να σας πω ότι έχω απόλυτη επίγνωση ότι αυτά τα επιτεύγματα, όλα όσα καταφέραμε στον τομέα αυτό, θα μπορούσαν να είναι βραχύβια αν αποδυναμωθεί αυτή η πολιτική βούληση. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να σας μεταφέρω. Θα πρέπει να εδραιωθούν τα αποτελέσματα και οι νέες ευκαιρίες που έχουμε διανοίξει τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια μπορούν τώρα να αξιοποιηθούν και να διευρυθούν, να αναβαθμιστούν. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ενότητα σκοπού, αποφασιστικότητα, πυγμή και πάνω απ' όλα πολιτική βούληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είχε ανέκαθεν νευραλγικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και οι ευρωβουλευτέ ήταν πολύ σημαντικοί παράγοντε τη εξωτερική μα πολιτική. Με τι διπλωματικέ μα αποστολέ, με τι αποστολέ παρατήρηση εκλογών, με την ε, Γενική Επισκόπηση των Πολιτικών μα, με ε, εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέλαβε τα μάλα στην Παγκόσμια Στρατηγική. Ευχαριστώ του προκατόχου σα και είμαι βεβαίω ότι και εσεί θα συνεχίσετε στην ίδια πορεία. Ο ρόλο σα λοιπόν είναι κέριος, είναι ρόλος κλειδί. Εσείς θα έχετε τον τελικό λόγο σε θεμελιώδη ζητήματα που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια. Θα έχετε τον τελικό λόγο για το νέο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα συμβάλλετε στη δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών για την εξωτερική μα πολιτική στο μέλλον. Οπότε η έκκληση που απευθύνω για μια ενωμένη Ευρώπη είναι ισχυρότερη σήμερα από ότι πριν από πέντε χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό να την ενισχύσουμε στο μέλλον. Η επιλογή της ευθύνη είναι δική σας και είμαι βεβαία ότι θα καταφέρετε να ανταποκριθείτε στο αίτημα αυτό, στην έκκληση αυτή, με τον πιο αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο και θα συνεχίζετε να, επενδύετε στον παγκόσμιο ρόλο της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, Αντιπρόεδρο και Πατή Εκπρόσωπη. Ξεκινάει τώρα ο γύρος των παρεμβάσεων των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, ο λόγος στον κύριο Γκάλερ. Για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για την εκλογή της κυρίας Φοντερ Λάιν. Είμαι πεπισμένος ότι ιδιαίτερα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας μαζί με τον Ζωζέ Μπορέλ και άλλους θα μπορέσει να υιοθετήσει σταθερές θέσεις. Όλοι θέλουμε σε ένα πολυμερές σύστημα να βασίσουμε την ε, διεθνή ε, τάξη και να εκπροσωπηθούμε από κοινού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή ήταν υπέρ της ε, υιοθέτησης αυτής της παγκόσμιας στρατηγικής και θα συνεχίσουμε και σε αυτή τη θητεία σε αυτή την πορεία. Για παράδειγμα, θέλουμε να υπάρξει το νέο μέσο NDICI να ε, δημιουργηθεί με τη δική μας επιρροή. Θεωρούμε ότι οι κρίσεις που υπάρχουν ε, κοντά μας και γενικότερα είτε στο νότο είτε στην ε, νοτιοανατολική μας γειτονία όλες αυτές οι κρίσεις καλούν για κοινή αντιμετώπιση και όντως έχουμε κοινά συμφέροντα και από αυτά τα κοινά συμφέροντα κανείς δεν μπορεί να διαχωρίσει τη θέση του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Πύρη, 1,5 λεπτό. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από τρία χρόνια το σώμα μας ε, χαιρέτησε την ε, ίδρυση της παγκόσμιας στρατηγικής για να έχουμε μια ισχυρή, ανθεκτική και συνεπή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξωτερική μας δράση ήθελε ένα πραγματιστικό όραμα που να καθορίζει σαφώ του στόχου μα, τα συμφέροντά μα, τα μέσα και φυσικά του εταίρου. Κάναμε πολλά έκτοτε. Γιατί υπάρχει ε, πρωτοφανής ε, παγκόσμια αστάθεια. Και γι' αυτό η παγκόσμια στρατηγική ενίσχυσε τι πολυμερεί εταιρικέ μα σχέσει και μα βοήθησε να συμμετάσχουμε περισσότερο στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Αξιόλογη πρόοδο έγινε σε μια σειρά από ασφάλεια και άμυνα πρώτα απ' όλα. Πρέπει να οικοδομήσουμε περαιτέρω γιατί έχουμε πολλά ζωτικά θέματα ενώπιόν μας. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρχει σαφής ενωσιακή προοπτική για τις ε, χώρες της διεύρυνσης. Δεύτερον, μια δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση της μετανάστευσης. Και τρίτον, ισχυρή συνεργασία με τις ε, χώρες στα σύνορά μας για ουσιαστική πολιτική γειτονία. Ναι, ο κόσμος ε, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από το 2016. Οι ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του κράτους δικαίου αφισβητούνται ακόμη και εντός μας. Και οι πλατφόρμες στις οποίες συμμετέχουν οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ε, αποσταθεροτυπτικές ε, επιπτώσεις και έχουμε και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό η Ευρώπη χρειάζεται τον κόσμο και ο κόσμος χρειάζεται την Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τις υπάρχουσες και τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις επιτυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για το Renew Europe η κυρία Φάουτμαντς. 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Μογκερίνη, όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν από τρία χρόνια, με τους εταίρους μας εκπονήσαμε αυτήν την ε, παγκόσμια στρατηγική. Τότε ήταν ζωτική σημασία. Το Κοινοβούλιο είχε καλέσει για κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό. Θέλαμε να έχουμε αυτή την πηξίδα για την εξωτερική μας δράση, για την εξωτερική μας δράση στον κόσμο. Και ήταν μια περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας. Με αυτή την ε, παγκόσμια στρατηγική έχουμε αυτό το μπούσουλα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στον κόσμο που να ξεκινάει από την ήπειρό μας και το είπατε κι εσείς σαφέστατα ότι όπου υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και Είχαμε λοιπόν αποτελέσματα για τα οποία μπορούμε, μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Πέσκο, άμυνα, οι διάφορε αποστολέ. Τι αναφέρατε πολύ σωστά. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Η διευκόλυνση για την ειρήνη επίση είναι ένα περαιτέρω βήμα. Δείξαμε ότι είμαστε αξιόπιστο εταίρο. Πολλοί μα κατηγορούν. Αλλά επιτύχαμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα και είναι σημαντικό να προσβλέπουμε και στο μέλλον. Τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε Πού πρέπει να εστιάσουμε. Και σήμερα νομίζω που έχουμε μια νέα πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φοντερ Λάιεν, και που είχαμε μια πολύ ενδιαφέρον συζήτηση μαζί της, δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε περισσότερα. Μπορούμε να έχουμε ισχυρότερη και πιο ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε προς ένα Ευρωπαϊκό στρατό. Και σας ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη Είχαμε πολλές καλές συζητήσεις, ε, πολλά βράδια σε αυτό το σώμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παγκόσμια στρατηγική σας αυτή. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Από τον κύριο Κλέρφοξ, τη δέχεστε. Ο κύριος Φόξ, παρακαλώ. Η κυρία Φόξ, συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω, εάν οι λαοί και οι δήμοι των διαφόρων κρατών ψήφισαν ποτέ ή ποτέ τους δίθηκε να ψηφίσουν για ένα ευρωπαϊκό στρατό. Αυτό είναι μια τεράστια ομοσπονδιακή επιβολή που είναι κατά της κυριαρχίας και της δημοκρατίας. Είναι ένα τρομακτικό μιλιταριστικό εγχείρημα ότι τολμά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προτείνει να έχει εξωτερική πολιτική. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση αν ζει σε ένα εθνικό κράτο να ελέγξει αυτού που ε, είναι αρμόδιοι για την κοινωνία σου για να δρουν υπεύθυνα στην εξωτερική πολιτική. Αλλά ότι το σώμα εδώ θα είχε το θράσο να ζητάει κάτι τέτοιο για το οποίο δεν έχει ψηφίσει κανεί είναι φοβερό αντιδημοκρατικό και φυσικά το κόμμα για τον Brexit δεν το στηρίζει. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Νομίζω ότι η μπλε κάρτα ήταν για να γίνει ερώτηση. Δεν άκουσα καμία ερώτηση. Ε, απλώς κάποιος είναι κατά του Ευρωπαϊκού Στρατού μας είπε. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου δείχνουν ότι ο λαός είναι υπέρ περισσότερης συνεργασίας στη, στα αμυντικά θέματα και εγώ προσωπικά είμαι υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Στρατού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ υπενθυμίζω ότι οι μπλε κάρτε είναι ακριβώς για να κάνετε ερώτηση ε, στον προηγούμενο μιλητή για να μπορέσει να απαντήσει. Και τώρα από πλευρά ε, των Πρασίνων ο κύριος Μπιτιχόφερ. δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Ιπατέ, εκπρόσωπε, αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ ενός ευρωπαϊκού στρατού και μεγαλύτερης συνεργασίας για την άμυνα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια παράπλευρη παρατήρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μία από τις πρώτες συζητήσεις σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι για την Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτό θα βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών εργασιών μας ε, στα επόμενα χρόνια και